έχει μείνει ένα θέμα σε εκκρεμότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας έχει γίνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομική κάλυψη των προγραμμάτων αυτών, αλλά η, η πρόβλεψη αυτή από ό,τι φαίνεται δεν επαρκεί Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη που υπάρχει να τριπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν, επαναλαμβάνω, οι πιστώσεις οι οποίες προορίζονται προς την κατεύθυνση της κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών. Τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αποκλίνει επιτέλους από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα. Το τελικό πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένες επενδύσεις και για την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας, η οποία θα πρέπει το 2020 να παράγει το 1 πέμπτο της απαιτούμενης ενέργειας. Όπως επίσης και την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, ηλιακής ενέργειας. τότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών μας και να μην εξαρτώμεθα πλέον από τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα το οποίο τίθεται τώρα είναι πώς θα μπορέσουμε όλες αυτές τις προβλέψεις να τις συγκεκριμενοποιήσουμε. Έχουν προβλεφθεί ε, αρκετές πιστώσεις και για το θέμα της συγκέντρωσης του άνθρακα έτσι ώστε να βρεθούν ε, λύσεις επιτέλους στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει και στην, ε, στη συνδυασμένη προσπάθεια του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα και γι' αυτό κάνουμε εργασίες ε, για την σωστή κατανομή των επενδυτικών προσπαθειών του επενδυτικού βάρους προβλέπονται προγράμματα τα οποία θα αποτελούνται κατά 70% από ιδιωτική χρηματοδότηση και κατά 30% από δημόσια και για τα προγράμματα υψηλού κινδύνου οι δημόσιες επενδύσεις φυσικά θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο κομμάτι. Θα πρέπει να καθορίσουμε εκ νέου το επίπεδο επενδυτικής ε, προσπάθειας και κάθε φορά που τα προγράμματα τα οποία έχουμε μπροστά μας προσθέτουν μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία, τότε θα πρέπει να, καλύψουμε, να τα καλύπτουμε οικονομικά. Προφανώς ε, βέβαια αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα δεν δίνουν λύση σε σχέση με τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Γι' αυτό και η κοινοβουλευτική μας επιτροπή έχει προσπαθήσει να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της χρηματοδότησης, για το οποίο επαναλαμβάνω υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά. Θα εξαρτηθεί το πώς θα πάνε τα πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίσει τις προτεραιότητες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μετά το 2020. Ένα δεύτερο θέμα είναι το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα επιπλέον δημοσιονομικά μέσα τα οποία μπορεί να έχει στη διάθεσή της μέσω μετακινήσεων από διαφορετικές θέσεις. ιδιαίτερα σχετικά με τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι από το 8ο πρόγραμμα δράσης. Και τέλος, τελευταίο θέμα, το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει και άλλες ε, τεχνολογικές μορφές παρέμβασης όπως το θέμα της συγκέντρωσης του άνθρακα όπως επίσης και της παραγωγής από εναλλακτικές μορφές ε, παραγωγής ενέργειας. Όλα αυτά τα θέματα δεν τα ακούτε για πρώτη φορά και τώρα πλέον το μόνο που ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Ρέγη και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου έχει το λόγο. Ε, Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω τη σημασία του στρατηγικού σχεδίου ενέργειας και τη συμβολή του για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καθαρών βιώσιμων μορφών ενέργειας και αποτελεσματικών. Χωρίς αυτό το σχέδιο αποκλείεται να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για το 2020. Ούτε πρόκειται να εξασφαλίσουμε την μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα που είναι στόχος για το 2020. Υπάρχει σύμπρια μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ανάγκη και τη σημασία και των στόχων του σχεδίου, αλλά και των μέσων με τα οποία θα πρέπει να το εφοδιάσουμε. Το Συμβούλιο Ενέργεια πρόκειται να εθετήσει κάποια συμπεράσματα για το SET Plan στη συνεδρίαση τη 12 η Μαρτίου την Παρασκευή δηλαδή. Και θα αποτελέσουν τα συμπεράσματα αυτά σημαντικό εφόδιο για το Συμβούλιο τη 25η Μαρτίου, γιατί οι κλιματικέ αλλαγέ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών αυτού του Συμβουλίου. Η χρηματοδότηση θα είναι τμήμα των συμπερασμάτων, αλλά με αρκετά συνετό τρόπο. Φυσικά δεν θα προεξοφλήσουμε και τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Τα πρωταρχικά στοιχεία της πρώτης συμπερασμάτων του Συμβουλίου είναι τα εξή. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από, τις από τα τεχνολογικά φύλλα στην επιχειρησιακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Αυτό να γίνει σταδιακά, προοδευτικά, αλλά με τον γρηγορότερο δυνατό ρυθμό και θέλουμε και μια συνεργασία ενεργειακή ε, και ερευνητική στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα εθνικά κονδύλια και να δημιουργήσουμε συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και συνεργασία της βιομηχανίας. Επίσης θέλουμε μια πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις, ε, όλους τους ενδιαφερόμενους Χρηματοπιστωτικού φορείς και ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών για να γίνει καλύτερος συντονισμός ε, των δράσεών τους. Επίσης, δεδομένη της ε, ε, εμβέλεια αυτής τη χρηματοδότησης από δημόσιο και ιδιωτικό κλάδο, θα πρέπει να προβλέψουμε αύξηση του μεριδίου κρατικής χρηματοδότησης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το λάβουμε δεόντως υπόψη και στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού αλλά και στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέταρτον, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρατηρηθούν και να ενθαρρυνθούν για να προσφέρουν κατάλληλα ενάψματα για να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική αυτή και αν χρειαστεί θα πρέπει να αυξηθεί και σημαντικά η χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό για την ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Πέμπτον, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζονται για να ε, βελτιώσουν το συντονισμό και τη συνέχεια της χρηματοδότησης τέτοιων ε, πειραματικών σχεδίων σε τομείς ενέργειας με υψηλό τεχνολογικό κίνδυνο. Επίσης, ε, ενεργοποιούν και κινητοποιούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης και ιδιωτικές και δημόσιες. Τέλος, η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αξιολογεί τα ε, βέλτιστα πακέτα χρηματοδότηση για μεγάλα σχέδια επίδειξη. Γι' αυτό και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τρόπου συνδυασμού πόρων από διάφορε πηγέ για να μπορέσουμε να περάσουμε και στην εμπορευματοποίηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν ένα απερίφραστο μήνυμα τη επένδυση που κάνουμε σε τεχνολογίε με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα παρά τι σημαντικέ ε, ε, δημοσιονομικές περικοπές. Ε, το μήνυμα του Συμβουλίου Ενέργειας της Παρασκευής θα είναι δέσμευση και ε, σημασία του θέματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, όλα τα κρατη θα πρέπει να επενδύσουν τέτοιες τεχνολογίες με χαμηλή χρυσή άνθρακα. Τώρα ο Επίτροπος, ο κ. Ποτότσικ, έχει το λόγο εξ της Επιτροπής. Thank you, President. Distinguished members of European Parliament, Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ συνάδελφο Ότιγκερ, αλλά με μεγάλη χαρά θα συζητήσω μαζί σας το θέμα των νέων τεχνολογιών. Έχω εμπλακεί από κοντά στο πρόγραμμα στρατηγικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών είναι θα έλεγα το θεμέλιο της πολιτικής την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση του Κοινοβουλίου του Ιουνίου του 2008 ήταν ξεκάθαρη. Προτείνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο στόχων και δεν θα πρέπει εμείς να χαμηλώσουμε το επίπεδο αυτό. Θέσατε τρεις ξεκάθαρες ερωτήσεις και θα δώσω απάντηση. Πρώτον, προτεραιότητά μας για το 2010 μέχρι το 2020 και η εκκίνηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωτοβουλειών. Αυτές οι έξι πρωτοβουλίες ταυτίζονται με τις ε, προσπάθειες τις οποίες έχουμε θέσει σε τομείς όπως η αιωλική ενέργεια, εναλλακτικέ πηγές γενικότερα ενέργειας. Έχουμε προωθήσει και την αποτελεσματικότητα της ενέργειας προωθώντας το πρόγραμμα Smart Cities έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη χρήση των ενεργειακά αποτελεσματικών τεχνολογιών στις πόλεις και στις αστικές περιφέρειες. Στο εσωτερικό αυτών των πρωτοβουλειών, σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους, έχει καθορίσει προγράμματα δράσης για την περίοδο 2010-2020 με συγκεκριμένους στόχους και με τις δραστηριότητες που προβλέπονται για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το 2010. Το 2011 θα ξεκινήσει μόνο το Smart Cities. Η επόμενη ερώτησή σας απαιτεί μια αποτελεσματική και ικανοποιητική δημοσιονομική κάλυψη για μετά το 2014 στα πλαίσια του συνδυασμού ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε 8 δις κατ' Σήμερα δαπανούμε 3 δις. Απαιτείται λοιπόν πολύ περισσότερα χρήματα για να καλυφθεί η περίοδος συνολικά το 2010-2020. Η γεφύρωση του κενού αυτού είναι ένα βασικό πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια η προσπάθεια θα πρέπει να συγκεντρωθεί στους τομείς όπου η παρέμβασή μας θα είναι αποτελεσματική. Να αποφύγουμε πρέπει τις επικαλύψεις και να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς όπου είναι πιο συγκεκριμένες. Προφανώς οι επενδύσεις δεν είναι αρκετές έτσι όπως προβλέπεται από το 7ο και 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπως επίσης και από την εμπορία των ρήπων τα οποία έχουν ήδη προσημειωθεί για χρήση στο πρόγραμμα συγκέντρωσης ε, των ε, ρήπων άνθρακα. Απαιτούνται περισσότερες συνεπώς προσπάθειες και από πλευράς του ιδιωτικού και από πλευράς του δημοσίου τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Θα είμαι λίγο ξεκάθαρος θα έλεγα, τα χρήματα θα έλθουν από αυτούς που τα διαθέτουν ουσιαστικά Ρωτήσατε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει και περαιτέρω τεχνολογικές λύσεις και προτάσεις ενεργειακές. Άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες θα αναφανούν μέσα στην επόμενη χρονική περίοδο και γι' αυτό το σύστημα θα πρέπει να παραμένει ευέλικτο. Όπως είπαμε ήδη, στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας για αποτελεσματική ενέργεια θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα Smart City το 2011. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες και μέσω του συστήματος SETIS, το οποίο αφορά την ε, συγκέντρωση και αποθήκευση ενέργειας και νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε τους κατάλληλους τομείς χρηματοδότησης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης της χρήσης της ε, εναλλακτικής πηγής ενέργειας στον τομέα της, ε, του κλιματισμού και της θέρμανσης και νομίζω ότι υποστηρίζονται όλες αυτές οι προστάσεις μας από όλους τους ενδιαφερομένους. Αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας, για την Ευρώπη, για το μέλλον. Τώρα θα πάρουν το λόγο μιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δύο λεπτά. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, με χαρά σας ξαναβλέπω εδώ, κύριε Πότοσνικ, στην ε, ε, στα καθήκοντά σας ως επιτρόπου για το Περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και θα ήθελα να απευθύνω ε, τα συγχαρητήρια μου στον Στέλφο Ρόιλ για την προφορική του ερώτηση και ευχαριστώ εσάς κύριε Επίτροπε για τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσετε τις την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, νέα τεχνολογία, στην τεχνολογία με χαμηλά ποσοστά άνθρακα. Φαίνεται ότι θα χρειαστούμε επιπλέον 40% ε, ενεργειακές πηγές για το 2030, από ό,τι προβλέπουν οι επιστήμονες, για την κατανάλωσή μας, η οποία θα αναπτυχθεί περισσότερο στα κράτη εκτός του ΩΣΑ. Και άρα το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνουμε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις για αναδίπλωση, για λιγότερη ανάπτυξη, για οτιδήποτε άλλο, αλλά θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια τα οποία ενδεχομένω προκαλούν και διχασμούς μέσα στις πολιτικές ομάδες, στα πυρηνικά δηλαδή ζήτηματα. Στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, όπου πολλά κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει αρκετά, χωρίς αυτό όμως να μας δίνει ιδιαίτερα προνόμια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μας υποχρεώνει όμως να συζητήσουμε σοβαρά την χρήση και την χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη χρηματοδότησή της, καθώς έχει, δεν έχει άνθρακα, δεν έχει εκπομπέ άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια. Και γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, θα θέλαμε και την υποστήριξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα καταθέσουμε τι σχετικέ τροπολογίε και θα ήθελα κλείνοντα να πω δύο λόγια για τα υποπροϊόντα τη πυρηνική ε, παραγωγή που απασχολούν ιδιαίτερα τον πολίτη. Υπάρχουν δύο λύσει, είτε η μακροχρόνια ε, αποθήκευση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ ω λύση, είτε η ανακύκλωση με την επαναξιοποίηση που ε, χρησιμοποιούν ως λύση η Γαλλία μαζί με τη Ρωσία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες ε, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι, αυτές είναι οι λύσεις τις οποίες μπορούμε να δώσουμε με τρόπο ευσυνείδητο και ενσυνείδητο. Ευχαριστώ πολύ. Των σοσιαλιστών, ε, η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε Ποτότσνικ. Όλοι έχουμε επίγνωση ότι ήδη αρχίζει και διαφαίνεται μια σαφή συνένεση γύρω από την ιδέα ότι όσο ε, ταχύτερα πραγματώσουμε μια πράσινη και οικολογική οικονομία, τόσο πιο γρήγορα θα εξέλθουμε από την κρίση. Οι διάφορε μελέτε υπολογίζουν ότι η προώθηση του στόχου του 20% ε, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια θα δώσει ευκαιρία σε 2,8 εκατομμύρια εργαζόμενους στον κλάδο αυτών των τεχνολογιών μέχρι το 2022. τρίτα των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα προέλθουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το κλειδί βρίσκεται στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, η ομάδα μου τάσεται υπέρ τριών σημαντικότερων στόχων. Καταρχήν μια πραγματική δέσμευση για να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το set plan. Δεν αρκεί να ομοδοποιήσουμε τα προγράμματα στήριξης που υπάρχουν. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε μετατρέψουμε το στόχο μας σε αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα σε ό,τι αφορά την, αποτελεσματική, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό υπό το πρίσμα της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών και της αναδιαπραγμάτευσης των δημοσιονομικών προοπτικών. Και αν θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που χρειάζεται η οικονομία μας για να εξέλθει από την κρίση, είναι ζωτική σημασία να προωθήσουμε τη φάση επίδειξης των καινοτόμων τεχνολογιών και να διευκολύνουμε την υιοθέτησή τους ε, και την εφαρμογή τους στην αγορά. Ε, για να δημιουργήσουμε πράσινες θέσεις απασχόλησης και οικολογικές χρειαζόμαστε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση για να, για να ενισχύσουμε τους, τις σχέσεις μεταξύ το, της παιδείας και της βιομηχανίας. Επίσης ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ε, πόλους αριστείας και να καλύψουμε τα κενά και τις αδυναμίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων, η κυρία Χαλ για δύο λεπτά επίσης. Πρόεδρε, Μπορούμε να ορίσουμε όσου στόχου θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, αλλά δεν θα μπορέσουμε να του επιτύχουμε, ιδιαίτερα του μακροπρόθεσμου του 2050, εάν δεν επενδύσουμε ε, με εμβάθυνση και σύστημα σε μια βιώσιμη και αηφόρο τεχνολογία χωρί άνθρακα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ναι, διατυπώνουν τι επικρίσεις του, γιατί δεν τηρούνται οι στόχοι μείωση των εκπομπών άνθρακα αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πλησιάζει καν αυτά τα ποσοστά. Και γι' αυτό μια ε, βιώσιμο, ένα βιώσιμο πρόγραμμα ε, για χαμηλής, ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακες τεχνολογίες δεν θα μπορέσει να προχωρήσει διότι δεν υπάρχουν οι επενδύσεις, δεν υπάρχει η επαρκής στήριξη αυτής της μετατροπής που βλέπω εγώ στη δική μου την εκλογική περιφέρεια να έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχει την υποστήριξη, τη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε τους απαραίτητους πόρους και τις επενδύσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και εντοπιστεί και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει πιο συγκεκριμένε απαντήσεις ιδιαίτερα για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που χρειαζόμαστε επιπλέον κάθε χρόνο όπως μας είπε μόλις τώρα ο Επίτροπος. Και εν τέλει, ναι, πρέπει να βελτιωθεί η ε, χρήση, η αποτελεσματικότητα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και ιδιαίτερα τη διασφάλιση διαχείρισή της. Μια αηφόρος όμως πυρηνική ενέργεια κατά την άποψη της ομάδας μου αποτελεί σχήμα οξύμορο. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέες πρωτοβουλίες. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων, ο κύριος Τόρμς έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά. Thank you, uh, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το set plan νομίζω ότι είναι μια καινή πρόταση γιατί δεν έχει εφοδιαστεί με τα κατάλληλα κονδύλια. Οπότε θα πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να εκταμιεύσουμε κάποια κονδύλια. Και το χειρότερο είναι ότι τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το CNR e 300, το σχέδιο ανάκαμψης και κάποια κονδύλια που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προορίζονται όλα αυτά τα κονδύλια περισσότερο για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που είναι λιγότερο αποτελεσματικές και που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Σήμερα λοιπόν στην αγορά, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2008 και το 2009, πάνω από το 70% όλων των επενδύσεων ε, αφιερώνονταν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αιωλική, βιομάζα, ηλιακή ενέργεια. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να καταρτίζουμε ένα set plan και να προσημειώνουμε κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ουσιαστικά δεν δίνουν κανένα μερίδιο στις ανανεώσιμες πηγές και αφιερώνουμε κάποια κονδύλια σε πυρηνική σχάση και δέσμευση άνθρακα. Κάτι που δεν αναφέρεται στο έγγραφο αυτό. Αλλά σίγουρα εκεί διοχετεύονται τα περισσότερα κοινοτικά κονδύλια. Το πρόβλημα είναι ότι εξαιτία ε, τη δράση ορισμένων λόμπι δεν έχουμε το θάρρο να θεσπίσουμε τι κατάλληλε προτεραιότητε. Ακόμη και η IA, η Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια, που δεν είναι και καμία θόα περιστερά, έχει σαφέστατε προτεραιότητε. 55% όλη τη μείωση ε, διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να προέρθει από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί εμείς δεν αφιερώνουμε ούτε ένα ευρώ στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο ανάκαμψη. 35% της μείωση του διοξιδίου του άνθρακα θα προέλθει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί μόνο το πολύ 10% από τη δέσμευση άνθρακα και 10% από τα πυρηνικά. Αυτά τα λέει ίδια η, ε, η Υπηρεσία ατομική Ενέργειας. Ακόμη και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολοιπόμαστε, υστερούμε σε σχέση με τις συστάσεις που δίνει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στις χώρες. Το πρώτο, είναι, το πρώτο ζητούμενο είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεύτερο, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, δηλαδή μείωση διοξιδίου του άνθρακα χωρί κίνδυνο και μετά οι υπόλοιπε τεχνολογίε. Εκ μέρου τη ε, ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, ο κύριο Τσίτσεστερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου με την αιμονή της αριστεράς του Κοινοβουλίου με την ατομική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο ψηφίσματα προς εξέταση σήμερα, τα οποία όμως έχουν πάρα πολλά κίνα μεταξύ τους. Η πυρηνική τεχνολογία είναι η μόνη αποδεδειγμένα επιτυχής τεχνολογία που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπομπή ρήπων στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα και το πετρέλαιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις άλλες μορφές ενέργειας. Περισσότερες από αυτές είναι σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι παραγωγής και δεν ξέρω αν έχουμε πετύχει πολλά σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από ε, εναλλακτικές μορφές. Είμαστε μεν φιλόδοξοι, ε, αλλά είμαστε και φιλόδοξοι και επιτυχείς στις αποτυχίες μας. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την πυρηνική ενέργεια. Ήδη καλύπτει η πυρηνική ενέργεια ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναγκών μας. Αν όμως προχωρήσουμε σε νέες μορφές τεχνολογίας και χρήσης της τεχνολογίας όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα χρειαστούμε περισσότερα. Φυσικά και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, και την αιωλική ενέργεια από τη Βόρεια Θάλασσα ή ακόμα και την ηλιακή ενέργεια από τη Σαχάρα. Αλλά όλα αυτά απαιτούν μαζικές επενδύσεις και εδώ είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Τώρα εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς η κυρία Ματίας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, μιλούμε εδώ για σημαντικές επενδύσεις ευρωπαϊκές στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πολύ σημαντικές οι προκλήσεις, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση. Και μάλιστα είναι μία από τις προκλήσεις που θα αποκτήσουν κεντρικό ρόλο, αλλά δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Γι' αυτό και θέλουμε αποσαφηνήσεις για το θέμα αυτό. Δεν λείπει μόνο διευκρίνηση ως προς τη χρηματοδότηση, λείπουν και πολιτικέ διευκρινήσει. Μιλούμε για αποτελεσματική αποδοτικότητα, πυρηνικά, δέσμευση άνθρακα, βιοκαύσιμα, ηλιακή ενέργεια και μιλούμε για πρόβλημα τη ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι ο φθηνότερο τρόπο για τη μείωση των εκπομπών. Υπάρχουν όμω και άλλε πολύ πιο φθηνέ ε, μορφέ για τη μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, η μείωση της ενεργειακή ενεργειακής κατανάλωσης, η ανακατανομή, η μικροδιαχείριση. Αυτές είναι πολύ πιο φθηνές μορφές ε, Εξοικονόμηση διοξιδίου του άνθρακα ή βελτίωση τη πρόσβασης στην ενέργεια ή επένδυση στι υποδομέ. Θέλουμε διευκρίνηση στη χρηματοδότηση και να πετύχουμε τη φθηνότερη λύση. Εκτό από την έλλειψη χρηματοδοτική και πολιτική διευκρίνηση λείπει και κάτι άλλο που κατά τη γνώμη μου είναι κέρια σημασία. Μιλούμε πολύ συχνά για τι συμπράξει ε, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, λες και ήταν πανάκια η λύση, η θαυματουργή για όλα τα προβλήματα. Δεν κατάλαβα από πού θα προέλθουν τα χρήματα όταν μιλάτε γενικά και όριστα για σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου. Όλες αυτές οι συμπράξεις και εταιρικέ σχέσεις που συστηματικά ιδιωτικου κλαδου ολες αυτες οι συμπράξει και εταιρικε σχέσει που συστηματικα αναφερονται για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι κάτι πολύ αβέβαιο και όριστο. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται τα κονδύλια. Οι συμπράξει θα πρέπει να είναι σαφής ποιος θα πληρώσει. Γιατί πολύ φοβόμαι ότι αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη τελικά είναι οι φορολογούμενοι και οι καταναλωτές. Θα πρέπει να δούμε από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα κονδύλια. Γιατί ο ιδιωτικός κλάδος κάνει επενδύσεις, αλλά και είναι λογικό να περιμένουν απόσβεση των επενδύσεων, αλλά δυστυχώ μονοπολούν τα κέρδη αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει συστηματικά να επιρρύπτουμε στις επερχόμενες γενές ε, το πλήρωμα των τιμολογίων της ενέργειας. Κατάλογο των ομιλητών, των γεγραμμένων ομιλητών. Ο κύριος Έχλερ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν συμφωνούμε όλοι ότι υποστηρίζουμε το σχέδιο αυτό και συμφωνούμε ως προς το περιεχόμενο, του στόχου του. Ωστόσο τα προβλήματα είναι διτά. Καταρχάς, εδώ έχουμε στο Κοινοβούλιο, όπως επεσήμανε ο κύριος Τουρμενσίδη, αδυναμία να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη και μόνο μια ιδεολογική συζήτηση αναπτύσσουμε σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Αυτό άλλωστε θα το δούμε και ως κύριο σημείο της σημερινή ψηφοφορίας. Δεν μπορέσαμε να βρούμε συμβαστική λύση για το σχέδιό μας έτσι ώστε να ορίζουμε τι είδους κριτήρια ορίζουμε. Κριτήρια όπως αηφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια προμηθειών. Γιατί θέλουμε μια ανοιχτή στις τεχνολογίες ε, προσέγγιση και να γίνει βεβαίως ιδεολογική αν θέλετε συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια αλλά αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι και η τελευταία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να επιτύχουμε εάν τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να τηρήσουν μία προσέγγιση συνεπή στην ενεργειακή τους πολιτική. Το Συμβούλιο έχει μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις ε, εξετάσει το ζήτημα λοιπόν δεν θα κρυθεί τόσο ως προς το προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος, αλλά ως προς την αντιπαράθεση δυνάμεων και την ε, βαρύτητα που θα δοθεί ε, στους διάφορους τομείς του σχεδίου μας, της, της ενεργειακής μας πολιτικής και το, κυρίως πού θα μπουν τα χρήματα, πού θα δοθούν τα περισσότερα χρήματα. Μπορούμε λοιπόν να ορίζουμε το ένα χρονοδιάγραμμα μετά το άλλο αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα. Δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε σε μια αντιπαράθεση απόψεων για τις λεπτομέρειες. Πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή πλέον να προχωρήσει την υλοποίηση. Τώρα το λόγο θα πάρει για ένα λεπτό η κυρία Σκόγκο. Ehm, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καλή πόθη, αλλά ανεπαρκής. Αν θέλουμε μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις έξυπνες πόλεις και όλα αυτά, χρειαζόμαστε και έξυπνες και μείζονες επενδύσεις. Έχουμε τα θέματα της θεμελιώδης έρευνας που απαιτούν μεγαλύτερη ανάμειξη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας στις πολιτικές μας προτεραιότητες και στους υψηλού μας στόχους. Μιλούμε για ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να θεσπίσουμε σαφώς τι προτεραιότητές μας και να κάνουμε μια ανακατανομή των κονδυλίων προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τους στόχου μα. Μόνο έτσι θα δώσουμε αξιοπιστία στο ΣΕΤ πλάν αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς μικρόφωνο. Thank you. It's years. Εδώ και τρία χρόνια έχει προσδιορίσει τους στόχους του το Συμβούλιο με 12 ε, σχέδια CCS τα οποία θα έπρεπε μέχρι το 2015 να έχουν, να έχουν φτάσει στην φάση της ε, ε, επίδειξε σχέδια για την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε το πώ θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια, αλλά μέχρι το τέλο του προσεχού μόνο χρόνου θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το σχέδιο το οποίο θα κρυθεί κατάλληλο για τη χρηματοδότηση. Αυτή το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ στενό λοιπόν, δεν έχουμε περιθώρια για να ικανοποιήσουμε τι προθεσμίε του 2015. Ε, γιατί διαρκώ έχουμε προβλήματα σε κάθε βήμα μα, κάποια ε, μικροπροβλήματα και ε, Ερωτώ λοιπόν εάν μπορούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε οι πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από το σχέδιο απόφασης να διατηρηθούν. Δεύτερον, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτροπολογίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει την ανακοίνωση της σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ε, δημόσια ανακοίνωση, έτσι ώστε, αν, έτσι ώστε να, να μπορέσουμε να τηρήσουμε το αυστηρό αυτό χρονοδιάγραμμα, να μην χάνουμε χρόνο. Και άλλο ένα παράγον καθυστέρηση ενδέχεται να είναι η διαδικασία καταθέση των, των ε, αιτήσεων από τους ενδιαφερομένου για τους αγωγού, για τον εξοπλισμό, το δίκτυο ολόκληρο για την αποθήκευση και δέσμευση του άνθρακα που ε, μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τελείως ε, το πρόγραμμά μας, τον προγραμματισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να αρχίσουμε τώρα τον προγραμματισμό αυτών και να αρχίσουν τα χρήματα να εισραίουν. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ζουμάνσκι θα πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, το ψήφισμα και ανακοίνωση πολύ σωστά δίνει έμφαση στην, ε, στις κλιματικές αλλαγές και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ε, ακούω πολλές ε, φωνές κατά της πυρηνικής ενέργειας. Και όμως είναι ο μόνος ε, τρόπος, που έχει, ο μόνος τρόπος ε, παραγωγής ενέργειας που έχει χαμηλό διοξείδιο το άνθρακα και κακώς ε, επικρίνεται τόσο δρυμαίος. Θα πρέπει να, να κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να λάβουμε υπόψη και την εμπορική τους απόδοση. Επίσης, μιλούμε για τη στρατηγική υλοποίηση μεγάλων ε, σχεδίων υποδομών και βελτίωση διασύνδεσης. Αυτή τη στιγμή όμως ε, έχουμε πρόβλημα στην ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα. Καλό. Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, ξέρουμε όλοι καλά ότι ένας ναρκωμανής μπορεί να είναι επικίνδυνος γιατί θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναβρει τη δόση του, για να εξασφαλίσει τη δόση του, την τόπα του. Και ξέρουμε ότι η αδίποτε μορφή εξάρτησης είναι ανεπιθύμητη, είναι κακό πράγμα. Πρέπει να την καταπολεμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει εξάρτηση οικονομική εξάρτηση όλο και μεγαλύτερη λόγω των εισαγωγών των πρώτων υλών για τη λειτουργία της οικονομίας μας. Πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξει. Οι επενδύσεις για τις νέες ε, ε, οικονομίες, για τις νέες ενέργειες, συγγνώμη, για την ηλιακή, για την αιωλική ενέργεια, για τη βιομάζα πρέπει να ενισχυθούν. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι με αυτές τις τεχνολογίες μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Εάν μάλιστα δεν επενδύσουμε σε αυτές, όλο και θα ενισχύεται η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και θα επιδεινώνεται διαρκώς η κατάσταση λόγω και της ρίκνωσης των σχετικών κοιτασμάτων ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εάν δεν κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, δεν θα μπορέσουμε ούτε και τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις να ε, ενισχύσουμε. Εκείνες οι οποίες χρειάζονται πραγματικά την ενίσχυσή μας, την υποστήριξή μας, ε, γιατί αποτελούν και το ζωτικό παράγοντα της κοινωνίας μας. Χρειάζεται επίσης να επενδύσουμε στις νέες αυτές τεχνολογίες προκειμένου να αντιπαρέλθουμε τα εμπόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή ως προς την εξισορρόπηση των δικτύων ε, μπορούμε να κάνουμε μεγάλο, καλό μείγμα τεχνολογίας με την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια και τις ε, νέες μορφές ώστε να μειώσουμε όλο και περισσότερο την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ε, στραφούν σε εκείνες τις τεχνολογίες όπου χρησιμοποιείται περισσότερο η ηλιακή, η αιωλική ενέργεια και η βιομάζα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Yes. Er Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την ε, πρόταση που κατατέθηκε και την πρόταση για ε, επενδύσει ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Τα δύο τρίτα των κονδυλίων από ό,τι αναφέρεται θα ε, αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών, την ηλιακή, την αιωλική, τη βιομάζα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα πρέπει να φροντίσουμε με τις νέες αυτές τεχνολογίες και να ξεπεράσουμε τη μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Μιλήσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδων νέες και οικολογικές θέσεις εργασίας χάρη στις νέες αυτές τεχνολογίες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαν στόχο την ανανεώσιμη τεχνολογία, την ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες δεσμεύσεις και τη χρηματοδότηση και ταυτόχρονα να, βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ήδη απασχολούνται στον τομέα αυτών, στον τομέα της ενέργειας δηλαδή, ώστε να καταρτιστεί, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, έχω δύο παρατηρήσει. Καταρχήν, είναι σημαντικέ οι επενδύσει σε τεχνολογίε χαμηλών εκπομπών άνθρακα και το θέμα τη δέσμευση άνθρακα στην γεωργία. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή τη στο τραγικό σχέδιο τεχνολογίες ενέργειας. Για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 χρειαζόμαστε πιο στοχοθετημένες και αυξημένε επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επίση θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε τις ε, κλιματικές αλλαγές. Εκεί η Γεωργία μπορεί να συμβάλλει στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020. Επίσης τα βιοκαύσιμα και η βιομάζα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ε, γεωργούς να μειώσουν τις εισαγωγές της. Τις τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα, τις δυνατότητες της γεωργίας και να αξιοποιήσουμε και τη γεωργική υγεία για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 επενδύοντας στη δέσμευση. Επίσης ε, το SET Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χαμηλές τεχνολογίες άνθρακα θα πρέπει να υποστηριχθεί. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία να συζητηθούν οι επενδύσει σε τεχνολογίε χαμηλού εκπομπών άνθρακα, αλλά ιδιαίτερω και στην ε, εξοικονόμηση ενέργεια και την ασφάλεια των προμηθειών. Και θα ήθελα να δω ιδιαίτερω πώ χρησιμοποιούνται τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμεί ήδη στη δική μου περιφέρεια έχουμε 250 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για οικονομική ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα, χαμηλή χρήση άνθρακα. Ωστόσο, η ε, επενδύσεις αυτές βλέπουμε ότι αποδίδουν ε, καλά, χωρίς όμως να έχουν ανέλθει στο επίπεδο που θα θέλαμε. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της έρευνας. Ήδη έχουμε ε, στην περιοχή μου υπογράψει μερικές εκατοντάδες συμβάσεις στην του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Ε, Ωστόσο τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και οι ανελαστικές δομές αποτρέπουν μερικές φορές τους ενδιαφερομένους. Είναι ε, φοβερές οι καθυστερήσεις ιδιαίτερα στην καταβολή των τελευταίων ποσών στους δικαιούχους. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να διδαχθούμε από το παρελθόν και να φροντίσουμε τα κονδύλια που θα αρχίσουμε τώρα να, να τα διαθέτουμε καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, σίγουρα χρειαζόμαστε μια στρατηγική μετάβαση τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βέλτιστη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Χάρη στι νέε ενέργειε μπορούμε να μειώσουμε κατά 17% τη χρήση ενέργεια στα κτίρια και κατά 20% στι μεταφορέ. Με έξυπνε τεχνολογίε ενέργεια μπορούμε να μειώσουμε κατά 10% τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Θα πρέπει επίση να βρούμε ένα σωστό τρόπο καταμέτρηση τη κατανάλωση ενέργεια και να βελτιστοποιήσουμε την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια χρήση ενέργεια. Για όλου αυτού του στόχου χρειαζόμαστε κάποιε κοινέ προδιαγραφέ και δίκτυα που θα εξασφαλίζουν διασύνδεση και διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σχέδια μεγάλη εμβέλεια για να χρησιμοποιήσει τι έξυπνε τεχνολογίε και τα έξυπνα δίκτυα και να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε αυτά των κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν δικές τους τέτοιες τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε ναύσματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επενδύσουν τέτοιες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών. Το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη και ευφυή βιομηχανική πολιτική που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα, τις θέσει εργασία και την παραγωγικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίε χαμηλών στον άνθρακα θα επιτρέψουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφύγει από την ε, μεγάλη κρίση και μπορεί να δημιουργήσουν μέχρι και 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε νέες ε, πρωτοβουλίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, θα πρέπει, ενέργειας και θα πρέπει τα σχέδια αυτά να τα ενσωματώσουμε και στο Ευρωπαϊκό Ηλεκτροδοτικό Δίκτυο και στις πράσινες μεταφορές και ε, σε άλλους αντίστοιχους τομείς. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε ευφύης πόλεις και σε ευφύή κτίρια, ιδιαίτερα σε κατοικίες. Και θα ήθελα να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός που, χωρί, που, αναγνωρίζει, που ε, προσδιορίζεται για, την, για τα εφή κτίρια, η κτίρια ε, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτός ο τομέας περισσότερο. Θέλουμε τουλάχιστον ένα 4% ποσοστό ε, μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την επένδυση στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μια συζήτηση προσαρμογής των ε, εθνικών οικονομιών στο στόχο της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε βέβαια επιχειρήματα και υπέρ και κατά των κλιματικών αλλαγών, γιατί δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι είναι ανθρωπογενείς οι αιτίες της, ε, των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό και θα πρέπει να προβληματιστούμε και να διαρωτηθούμε πώς θα εξασφαλίσουμε πόρους για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι διατάξεις για την έρευνα θα πρέπει να είναι πιο ελαστικές και να εξασφαλίζουν ε, τη χρηματοδότηση σε δυναμικούς ε, ερευνητές. Πώς θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς ε, υποστήριξης επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ τη ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά αυτό θα πρέπει, αυτά τα κονδύλια να εξασφαλιστούν ει βάρος της πολιτικής συνοχής. Κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23 Ιανουαρίου του 2008 για την υποστήριξη σε πρόωρο στάδιο των σχεδίων επίδειξης σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που είναι τμήμα του περιβαλλοντικού και κλιματικού πακέτου, ευρω... καταλήγει σε ένα set plan με διάφορα σχέδια επίδειξης. Το δικό μας ψήφισμα ασχολείται με το θέμα αυτό και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυστυχώς δεν είναι επαρκή για να υλοποιήσουν τους στόχους και να δημιουργηθούν τουλάχιστον 200 εγκαταστάσεις σχεδίων επίδειξης μέχρι το 2015. Το σημείο 18 αναφέρει ότι είναι απολύτως απαραίτητο τουλάχιστον 12 ε, τέτοιες εγκαταστάσεις ε, επίδειξης για τις οποίες χρειάζονται επενδύσεις να συνδυάζουν τρεις ε, διαφορετικές τεχνολογίες. Επίσης έχουμε 300, 300 εκατομμύρια άδειε για τις ε, εκπομπέ άνθρακα. Οι επενδύσεις στα σχέδια επίδειξη ε, θα εξαρτηθούν από τις ε, τιμές που επικρατούν στην αγορά. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υποστήριξη της καθαρής τεχνολογίας αφορά κυρίως έξι ε, σχέδια και δύο βιομηχανίες. Πώς το, το Συμβούλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποστηρίξει τη δημιουργία δύο ακόμη έως τεσσάρων τέτοιων εγκαταστάσεων επίδειξης. Είναι η εγγεγραμμένη ομιλήτρια κυρία Χέτσκοκ, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα, οπότε το λόγο θα πάρει ο κύριος Χέλμερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ακούσαμε πολλές ανοησίες σήμερα για πράσινες θέσεις εργασίας. Γεγονός είναι ότι η μονομανία μας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη πιέζει προς τα άνω τις ενεργειακές πηγές τιμές και ε, πιέζει ιδιαίτερα το πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη. Θα εγκαταλείψουν τελικά όλες αυτές τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και θα φύγουν για, πιο χαρμόσυνους ουρανούς και πάνω απ' όλα χώρους ανάπτυξη των, εργασιών τους. Αυτό θα σημάνει μεγάλο κόστος της ε, θέσης εργασίας. Μόνο μία μελέτη είδα από την Ισπανία για τις πράσινες θέσεις εργασίας, οποία επέδειξε ότι κάθε θέση εργασία στον πράσινο τομέα σημαίνει ότι χάνονται 2,2 θέσει εργασία από άλλον τομέα. Εάν θέλουμε λοιπόν με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, λύση είναι μόνο μία, είναι η πυρηνική ενέργεια. Έχουμε αρχίσει να συζητούμε τι νέε πυρηνικέ ικανότητε και αυτό είναι θετικό. Εάν θέλουμε λοιπόν να παραμείνει αναμένο το φω, χρειαζόμαστε μια πυρηνική αναγέννηση και τη χρειαζόμαστε τώρα. πολύ, κύριε Τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Καρβάλιο θα πάρει το λόγο. E η έρευνα και η τεχνολογία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας με χαμηλή χρήση άνθρακα. Θα πρέπει να ευνοήσουμε την μετάβαση σε μια τέτοια κοινωνία με έξυπνε πόλει, με αποκεντρωμένη διαχείριση ενέργεια και ανταγωνιστική οικονομία. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική, απαραίτητη προπόθεση για μια ευήμερη και βιώσιμη κοινωνία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ενεργειακό ανεφοδιασμό, να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ και να πρωτοστατήσουμε παγκοσμίω τη χρήση καθαρών ε, τεχνολογιών ενέργεια. Χαίρομαι με του βασικού προσανατολισμού τη ε, ανακοίνωση και την λογική της σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνδυασμό του κοινοτικού, εθνικού και περιφερειακού Προπολογισμού. Φυσικά χρειαζόμαστε αύξηση των δημόσιων κονδυλίων στην έρευνα για τις ε, καθαρέ τεχνολογίε. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει για την αύξηση και των ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο αυτό. Θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 8ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, τεχνολογική ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια, στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και στην προστασία του περιβάλλοντο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη της βιομηχανίας να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Η κυρία έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή δεν είναι μια συζήτηση τυπική και επίσημη. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη και να θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις τι πόρους χρειαζόμεθα, από πού θα πάρουμε τους πόρους αυτούς. Ελπίζω οι απαντήσεις να είναι πιο συγκεκριμένες και από την Επιτροπή και από το επόμενο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηκώσει πρώτη στον κόσμο της καταπολέμησης της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της κλιματολογικής πρόκλησης. Πρέπει να φανεί συνεκτική με τις επιλογές της αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αλλιώς θα τρωθεί η αξιοπιστία της. Όταν μιλάμε για οικονομία χαμηλών εκπομπών, σημαίνει μια ουσιαστική επανάσταση για το παραγωγικό μας σύστημα, για το βιομηχανικό σύστημα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους πόρους. Αυτή η επανάσταση του τύπου του Κοπέρνικου είναι απαραίτητη εφόσον θέλουμε να μείνουμε ανταγωνιστική. Σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια υπάρχει φαιά ουσία, υπάρχει επιθυμία, υπάρχει ικανότητα. Πρέπει και εμείς να παίξουμε το δικό μας ρόλο. Και η Επιτροπή και εμείς και τα κράτη-μέλη και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να συνδυαστούμε όλοι για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους της. Τώρα για Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι το πρώτο βήμα ο πρώτο κρίκο στην αλυσίδα είναι καλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση τη ενέργεια. Όμω θα ήθελα εγώ να επισημάνω την πολιτική σύγχυση και το άγχο το οποίο είναι διαδεδομένο προ τη χρήση τη βιοενέργεια βλέπουμε ότι αποφεύγουν πολλοί από τους συναδέλφους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της βιοενέργειας. Ιδιαίτερα όταν είχαμε προβλήματα ως προς τις τιμές των τροφίμων. Λίγοι ήμασταν εκείνοι οι οποίοι μιλούσαμε για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι γεωργία, οι περισσότεροι γεωργοί στην Ευρώπη. Τώρα με την έλλειψη εμπιστοσύνης και το πεποίθηση που αντιμετωπίζουν διότι έχουν πέσει τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν τη γη του για την ε, καλλιέργεια βιοκαλλιεργιών, για τις βιοκαλλιέργειες. Αυτό όμως στην Ιρλανδία δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια βεβαιότητα, βεβαιότητα την οποία πρέπει να μας προσφέρουν οι πολιτικοί με τις επιλογές τους. Ήδη την, την ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας τη βλέπουμε ορατή. Αλλά χρειάζονται κατάλληλες πολιτικές επιλογές. Διαφορετικά χάνουμε το χρόνο μας. ο κύριο Σταμπάτσου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τα στοιχεία που μας έδωσε. Στην περίπτωση των νέων κρατών μελών είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις πράσινες τεχνολογίες και το πέρασμα σε αυτές τις τεχνολογίες. Μια σημαντική δυνατότητα χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι τα λεγόμενα μεικτά συστήματα, όπως επίσης και το σύστημα εμπορίας ρήπων. Είναι μια καλή ευκαιρία για την κεντρική Ευρώπη και για τις βαλτικές χώρες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τους πόρους μας. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα μετά για να καλύψει τις δικές μας ανάγκες και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις νέες χώρες έτσι ώστε οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε να γίνουν αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης. Κατανοώ βεβαίω ότι οι νέες τεχνολογίες κοστίζουν πάρα πολύ. Το κατανοώ πλήρω αυτό. Σε σχέση τώρα με την κοινή αγροτική πολιτική θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με νέα μέτρα για αλλαγές στην παραγωγή, για νέους τύπους ζωοτροφών, για νέους τύπους μορφής εκμετάλλευσης των αποβλήτων κτλ. Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες ε, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ένωσης θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας καινοτόμας οικονομίας ε, με τη μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό σύστημα που θα ευνοεί τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σε σχέση με τις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα. Βέβαια, η, τα ορυκτά καύσιμα είναι μέχρι στιγμής ε, σημαντική παράδοση της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, σωστή μετάβαση και η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη δημιουργήθηκε χάρη στη χρήση άνθρακα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χρήση άνθρακα αυτή που τόσα χρόνια παράδοση έχουμε στην Ευρώπη από τη μια στιγμή στην άλλη. Βέβαια, η ενεργειακή πολιτική είναι σημαντικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η έμφαση που δίνεται σε αυτή είναι ένα καλό βήμα ε, για την ενίσχυση μιας καινοτόμας οικονομίας, αρκεί να λάβουμε υπόψη τη χρηματοδότηση της τεχνολογίας καθαρού άνθρακα. Αν θέλουμε να ελοπίσουμε τους φιλόδοξους στόχους μείωσης άνθρακα, θα πρέπει να επενδύσουμε στις έρευνες, σε καθαρές τεχνολογίες, σε ισορροπημένες τεχνολογίες και αποδοτικές. Επίσης, θα πρέπει να συνδυαστούν ε, οι πηγές από το δημόσιο και τον ιδιωτικό κλάδο γιατί πραγματικά η τεχνολογία μπορεί με βιώσιμο τρόπο να τροποποιήσει τη ζωή μας. Θα πρέπει όμως να τροποποιηθεί και ο τρόπος παραγωγής ενέργειας. Οι επενδύσεις σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα γίνουν μόνο όταν η κοινωνία βεβαιωθεί για τα δαψιλή κονδύλια που θα πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στρατηγικούς στόχους Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα πλαίσια της συζήτησης για τις ενεργειακές επιλογές υπάρχει μία βεβαιότητα. Ο πιο σημαντικός και φθηνός πόρος, ενεργειακός και αηφόρος είναι η ενέργεια την οποία συλλέγουμε, η σωρευμένη ενέργεια. Οι ορεινές περιοχές για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους είναι πρότυπο για την κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολύ χαμηλό επίπεδο άνθρακα. Παράγουν οι ορεινές περιοχές το σύνολο της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η περιοχή από όπου προέρχομαι στην Ιταλία παράγει το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στις ορεινές περιοχές υπάρχει σορευμένη εμπειρία και στην κατασκευή κατοικιών ιδιαίτερα αποτελεσματικών ενεργειακά χτίζουμε κτίρια τα οποία είναι επαρκή και σε επίπεδο ηλεκτρισμού και σε επίπεδο θέρμανσης, κατοικίες οι οποίες πολλές φορές παράγουν περισσότερη ενέργεια από όσοι καταναλώνουν με φυσικά χρήση προχωρημένων τεχνολογιών. Είναι θα έλεγα πρότυπα οι ορεινές περιοχές και για άλλες χρήσεις όπως η γεωθερμία, οι συσσωρευτές, η γεωθερμική ενέργεια και τα συστήματα διανομής. Οι ορεινές περιοχές έχουν ενέργεια, καθαρή ενέργεια και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να έρθει σε επαφή με τις ορεινές περιοχές, να τις εντάξει στη στρατηγική τους, να αναγνωρίσει το δικαίωμά τους σε αποζημιώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές τις οποίες παρέχουν ήδη. Το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζει τον ειδικό ρόλο των ορεινών περιοχών και γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρωτοβουλία για τη σωστή εφαρμογή του 174 και για μια σωστή πολιτική στον τομέα των ορεινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενέργεια. Δέχουμε έχουμε την έκθεση Duren Vargel της Επιτροπής Περιφερειών για τη συνεισφορά των ορεινών περιοχών στην ενεργειακή προβληματική σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών και σε επίπεδο ε, κατασκευών. Οι ορεινές περιοχές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της έκτασης της Ευρώπης ε, και 90 εκατομμύρια κατοίκους. Θεωρούνται μέχρι τώρα μη ευνοημένες περιοχές. Παρόλα αυτά ακολουθούν καινοτόμε πολιτικές και μπορούν να προλάβουν τη στέρησή τους, την ειστέρησή τους, με νέε παραγωγικές μεθόδους στα πλαίσια τη στρατηγική 20 20-20-20 αποδεικνύοντας ότι η αυτάρκεια ενεργειακή είναι πιθανή με σαφέστατα αναλήψιμο κόστος. Σε έχουν ζητήσει το λόγο οκτώ συνάδελφοι. Σας παρακαλώ κρατήστε το χρόνο του ενός λεπτού παρέμβασης για όλους. Ε, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Νικολέσκου. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συχνά κατηγορούμε την ε, γεωργία της Ευρώπης για την, ως υπέτεια για την ε, αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, πράγμα όμως το οποίο δεν ευσταθεί. Αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε το γεγονός ότι συμβάλλει το όντι σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα η γεωργία. Η δέσμευση λοιπόν και πεθήκευση άνθρακα, η βιομάζα είναι μέσα, πιστεύω, στα οποία θα μπορούσε να συμπράξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και η γεωργία. Έτσι όταν μιλούμε για τεχνολογία χωρίς άνθρακα θα πρέπει προτεραιότητα να αποτελεί η γεωργία και όχι το, το φτωχό συγγενή όπως έχει γίνει στο παρελθόν στην προηγούμενη στρατηγική για το 2020. Τώρα θα πάρει ο κύριος Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ δύο ονόματος, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να πω στον συνάδελφο εκεί απέναντι ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι διέξοδος και πάνω απ' όλα δεν είναι ανανεώσιμη πηγή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα είναι ωφέλιμα για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα, ναι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει αυτή η μείωση να μην επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθήσουμε τα μέτρα τα οποία θα προωθήσουμε, τα μέτρα στα οποία θα επενδύσουμε, έτσι ώστε να μην ε, μειώνουμε τις εκπομπές του άνθρακα από τη μία και από την άλλη να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας. Το 2010 ως έτος ε, βιοπικιλότητας νομίζω μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σύμβολο. Πρέπει να τηρήσουμε αυτό το στόχο. Όλες οι επενδύσεις, όλα τα μέτρα που θα αναπτύξουμε να έχουν σαν στόχο την αηφορία στο περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος μας και την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Πέρα θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η συζήτηση για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή εκπομπή άνθρακα θα πρέπει να μας απομακρύνει από το εξή γεγονός. Πολύ δύσκολα θα γίνουν άλματα αν ε, δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα ε, της εξάντλησης των βασικών πηγών ενέργειας, γιατί εμείς εξαρτώμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Και τα ρηκτά αυτά καύσιμα είναι πρώτη ύλη σημαντικότητα των βιομηχανιών, όπως είναι η χημική βιομηχανία και η φαρμακευτική βιομηχανία. Τα κοιτάσματα πετρελαίου που υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα θα πρέπει να ε, τα διαχειριζόμαστε με σοφία και σύνεση και με μεγάλη λιτότητα και με φιδωλό τρόπο. Επίσης, ε, το πρωτόκολλο του Σουψάλλας του 2002 και της Λισαβόνας του 2005 με πορίσματα επιστημονικά που μιλούν για την εχμή του πετρελαίου και την ε, σταδιακή μείωση των κοιτασμάτων πετρελαίου μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου γιατί αρχίζουν και σπανίζουν οι πόροι. Είναι λοιπόν λογικό να περνούμε σε άλλες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή πρέπει πιστεύω να ομολογήσουμε ότι δεν έχει χορηγηθεί απαραίτητη προσοχή στην πυρηνική ενέργεια μέσα στην έκθεση αυτή. Η λύσεις με τις αναλλακτικές πηγές, τη βιομάζα, την ηλιακή, την αιωλική ενέργεια, είναι λύσεις μακροπρόθεσμες και δεν θα μπορέσουν πάντα ίσως να μας δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να δράσουμε πολύ γρήγορα γιατί αν κοιτάξουμε και ότι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, την κρίση σχετική με το φυσικό αέριο, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, η πυρηνική ενέργεια είναι μια μεγάλη και σημαντική πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη μας προσφέρει πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού και θα πρέπει να την αναπτύξουμε κατά τρόπον ασφαλή. Είναι όρος εκτελώνουν κάνευ αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλλη έχει το λόγο. Äh, äh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και πρέπει να δούμε τώρα ε, τα ειδικότερα στοιχεία, πώς θα διατεθούν τα κονδύλια και πού θα εντοπιστούν ιδιαίτερα οι Ερευνητικέ προσπάθειε. Τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, συναντηθούν, να συζητήσουν οι πραγματογνώμων, οι από τα τρία θεσμικά όργανα, να ορίσουν μια ε, ομάδα μελέτης που θα προσδιορίζει και στόχους για τα κράτη-μέλη και θα μπορεί μετά να παρακολουθεί και να επιτηρεί τις δραστηριότητες έρευνας. Χρειάζεται να έχουμε όχι μόνο R&D, έρευνα και ανάπτυξη, αλλά R&D, δηλαδή έρευνα, ανάπτυξη και αποτελέσματα. Έτσι θα έχουμε ε, με το συντονισμό τα πιο καλά αποτελέσματα. Κύριε Κέλλη, θέλω να ρωτήσω την διερμηνία έχει αποκατασταθεί μετάδοση στα αγγλικά. Είχαμε αγγλικά, ήταν όλα εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μπάλτσκο. Elnök asszony, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν όλο καλά λόγια για τη μείωση των ρήπων, για τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν μας είπαν για την ουσία. Τα χρήματα, πού θα τα βρούμε. Υπάρχουν κάποιοι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, θα τους εκμεταλλευτούμε πλήρως. Αν δούμε τις προηγούμενες χώρες που ονομάζαμε σοσιαλιστικές, έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες και μπορούμε η στάση την οποία κρατήσαμε ε, στην Κοπενχάγη να πούμε ότι μας κάνει υπερήφανους. Μήπως μπορούν να πουλήσουν λοιπόν τις ποσοστώσεις τους για τις εκπομπές άνθρακα ε, και δεν θα πρέπει κανείς να αντισταματήσει. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας μιλάμε για δις ε, διαθέσιμα ουγγρικά φιωρίνια τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για όλους. Εφόσον θέλουμε λοιπόν πράσινες επενδύσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τους διαθώσιμους πόρους. Μέχρι τώρα τα αιτήματα της Ουγγαρίας δεν έχουν γίνει πλήρως δεκτά. Ευχαριστώ. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ο στόχος για το 2020 είναι χρήση κατά 20% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βέβαια για τη Ρουμανία ο στόχος αυτός είναι ακόμη πιο φιλόδοξος, ανέρχεται στο 24% με βάση κάποιες μελέτες. Και μάλιστα μια περιοχή στο νότια Ρουμανία χρησιμοποιεί ολική ενέργεια σχεδόν τόσο όσο και η Γερμανία. Είναι δεύτερη σε ένα κατάλογο επιδόσεων. Επίσης έχουμε το σημαντικότερο αιωλικό πάρκο με 240 ανεμογεννήτριες που θα παράγουν 600 και μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μάλιστα αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο θα ολοκληρωθεί φέτος και οι πρώτες 139 ανεμογεννήτριες θα αρχίσουν να λειτουργούν και μάλιστα και στην Κομιτεία της Κωνσταντζα θα έχουμε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Το σχέδιο αυτό είναι τεράστια σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ρουμανίας γιατί θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις ενεργειακές μας εισαγωγές. Grazie ε, Έχω την εντύπωση ότι σε δύο σημεία μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε πλήρως μετά από αυτά που ακούσαμε το πρωί. Εξοικονόμηση, αποτελεσματικότητα και ανανεούμενες πηγές ενέργειας. Δεν είναι επαρκές όμως το επίπεδο αυτό συμφωνίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε και σε άλλα δύο θέματα. Το πρώτο είναι η πυρηνική ενέργεια. Η λέξη πυρηνικός μας, κάνει, μας δημιουργεί αισθήματα φόβου. Ας προσπαθήσουμε να μην είμαστε συναισθηματικοί εδώ. Δεύτερον, η χρηματοδότηση μας, ε, κάποιες μορφές χρηματοδότησης ε, μικτής μας κάνουν να φοβόμαστε του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ιδέα ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε κοινέ πρωτοβουλίες με το δημόσιο ιδιωτικό χώρο είναι κάτι το οποίο πολλούς φοβίζει. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση. Δεν είναι σοβαρό ο δημόσιος τομέας να μην έρχεται σε επαφή και να μην συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται και το δημόσιο με τρόπο που σκέφτονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κύριο κύριος Σέχλερ παρενέβη σήμερα στη συζήτηση, αλλά θέλει να κάνει μια συμπληρωματική παρέμβαση. Σύντομα κύριε Έχλερ, σας παρακαλώ. Yes, please. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Βεβαίω έχουμε κάνει τη συζήτηση πολλέ φορέ. Είναι θεμητό να γίνουν ιδεολογικέ αντιπαραθέσει μεταξύ των ομάδων. Αλλά θα ήθελα να τυπώσω συγκεκριμένα την ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μου δώσουν απαντήσει. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν το χρονοδιάγραμμα. Ω προ τη χρηματοδότηση, ω προ την εφαρμογή, τι σκοπεύετε να κάνετε, ω προ την εφαρμογή του, το χρονοδιάγραμμα και οι προοπτικέ για τα κράτη-μέλη. Σύντομα, σα παρακαλώ. Ε. Äh, Δεν θα αναφερθώ στο ιδεολογικό ζήτημα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα τραβήξει μάκρο μια τέτοια συζήτηση, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Δύο συγκεκριμένα μέσα τα οποία θα δούμε την επόμενη εβδομάδα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, ότι από το Resharing ε, Finance Facility ε, βλέπουμε ότι περισσεύουν χρήματα. Αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και μου λένε ότι η Επιτροπή είναι εκείνη, η Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα δηλαδή, είναι εκείνη η οποία αποτρέπει τη διάθεση των κονδυλίων αυτών, την αποδέσμευσή τους υπέρ της ενέργειας. Δεν θέλει να θέσει αυτά τα κονδύλια στην δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα κτλ. Σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα μπορείτε να απαντήσετε κύριε Επίτροπε. Και δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον 15% των κονδυλίων από το recovery package, από την ε, δέσμη ανάκαμψης, περισσεύουν. Αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχουμε πει εμείς στο Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα για τα smart cities, για τις ευφυείς πόλεις. Μπορείτε να μου δώσετε και σε αυτό μια απάντηση. Τελευταία παρέμβαση σύντομη του κυρίου Ματούλα. Και μετά θα πάρουν το λόγο το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Κύριε Ματούλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει η χώρα μια συζήτηση για τις επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Κάτι που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πρωτοστατήσει παγκοσμίω στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών και να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Προσβλέπουμε σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα καθαρό περιβάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιες λύσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους της. Ας μην ξεχνούμε το τεράστιο δυναμικό της πράσινης οικονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατάγομαι από μια περιοχή της Ρουμανίας που έχει σημαντικότατο γεωθερμικό δυναμικό που δυστυχώς ε, δεν αξιοποιείται δεόντως μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να δώσουμε πιο κεντρικό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να ενθαρρύνουμε τις τοπικές αρχές να προωθήσουν τέτοιες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου. Έχει ο κύριος ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο σημείωσε προσεκτικά τις παρατηρήσεις ε, της πρωινής συζήτηση και σε μεγάλο βαθμό εστερνιζόμαστε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα τα συμπεράσματα που θετήσουμε αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Βιομηχανίας θα δημιουργήσουν μια πάγια βάση, θα διασκεδάσουν πολλές ανησυχίες και θα δώσουν ένα αρκτήριο λάκτισμα για τις ε, βιομηχανικές πρωτοβουλίες. Για αυτές τις πρωτοβουλίες υπάρχει συνένεση ότι θα έχουν κέριο ρόλο για τη μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης, για τη βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και θα δώσουν μια τεχνολογική όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απαραίτητες και για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Υπάρχουν και άλλες μελέτες, σας διαβεβαίω, πέραν αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταδεικνύουν τη θετική συνέπεια που θα έχει μια τέτοια επένδυση στην απασχόληση μέσω και μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα πλέγμα αρχών και κοινών πρακτικών για, για την ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλειών. Βέβαια θα πρέπει να προσδιορίσουμε και τα οικονομικά μέσα, τους πόρους και κάποια κριτήρια κρατικής παρέμβασης που θα ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών και το θέμα το οικονομικό. Επιμείνατε ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση. Την ανησυχία αυτή την συμμερίζεται και το Συμβούλιο. Βέβαια, δεν μπορούμε να σφετεριστούμε το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Θα ισχύσουν οι διατάξει περί χρηματοδότηση, αλλά όλοι επιμείναμε στην ανάγκη αύξηση του προπολογισμού για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών και το θέμα των προτεραιοτήτων, τη θέσπης προτεραιοτήτων θα αποτελέσει το επίκεντρο των μελλοντικών συζητήσεων σε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα της ασφάλειας ε, είναι σημαντικό και το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ε, την επαρκή χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών του σχεδίου ΣΕΤ και στο ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και στο επόμενο. Επίσης ε, θα ήθελα και εγώ να υπενθυμίσω όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γενικώ οι, οι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και η ιδιωτική χρηματοδότηση το ίδιο. Και εκεί θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά, ώστε ο αντίκτυπος των κρατικών κονδυλίων να βελτιστοποιηθεί και να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Για να τεθούν επιτυχώς ε, σε ισχύ αυτές οι πολύ σημαντικές ε, πρωτοβουλίες για το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Mr. Commissioner. Thank you. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προτάσεις σας. Παρακολούθησα τη συζήτηση από πολύ κοντά και υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μικρή περιγραφή, μια μικρή ιστορία. Μετά από την πετρελαϊκή κρίση του 70, Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σεβόμενοι το περιβάλλον και αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο ε, θα έλεγα εύρος. Αλλά οι προσπάθειες αυτές ε, και οι επενδύσεις τις οποίες κάναμε στις οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες ε, εξαφανίστηκαν ουσιαστικά γιατί έμειναν χαμηλές οι τιμές του πετρελαίου για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μια περίοδος ψευδέστησης, θα έλεγα για όλους, σχετικά με το αηφόρο της προσπάθειάς μας. και οι επενδύσεις τις οποίες κάναμε τότε μετά την πετρελαϊκή κρίση ήταν τετραπλάσιες σχετικά με αυτές τις οποίες διαθέτουμε σήμερα. Δεν φανήκαμε λοιπόν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν έπρεπε και δεν, μπορούσα, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της εξάρτησης από συγκεκριμένες μορφές ενέργειας. Πρέπει να προβλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Το να προβλέπουμε καλύτερα δεν σημαίνει ότι είμαστε ονειροπόλοι, σημαίνει ότι είμαστε πραγματιστές. Και αυτό ακριβώς και η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην πράσινη ανάπτυξη. Απαιτείται να έχουμε όχι να, να κάνουμε τις ε, βιομηχανίες μας πιο καθαρές, αλλά απαιτείται να είναι πλέον ε, συγκεκριμένα καθαρές οι βιομηχανίες και η παραγωγή μας, εφόσον θέλουμε και οι επενδύσεις μας να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, κάτι το οποίο είναι στόχος ε, της Ατζέντα 2020. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα, όλες οι προβλέψεις οι οποίες προβλέπονται για τις άμεσες επενδύσεις βασίζονται στα λεγόμενα roadmaps, στου οδικούς χάρτες. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αν εξετάσετε προσεκτικά τις προτάσεις οι οποίες γίνονται, πώς υπολογίζουμε τις ανάγκες, πώς προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες, θα δείτε ότι και στο Solar 16 θα δείτε ότι υπολογίζουμε συγκεκριμένα ποσά για, όλες, για όλα τα προγράμματα όπως το Smart Cities, τα νέα αποτελεσματικά συστήματα διανομής. Και έχουμε ένα συνολικό δίκτυο 75 και το 75 αυτό ε, από το 75 αυτό μόνο 7 είναι για την πυρηνική ενέργεια. Η ε, πυρηνική σχάση φυσικά δεν περιλαμβάνεται εδώ. Βλέπουμε ότι είναι σαφής ο προσανατολισμός της επενδυτικής μας προσπάθειας. Το θέμα είναι από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα χρήματα. Σας είπα το πρόγραμμα που έχουμε ε, ήδη προβλέψει μέσα από τους λεγόμενους οδικούς χάρτες. Χρήματα θα προέλθουν και από τη βιομηχανία και από τις οικονομίες ε, των κρατών μελών και από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις ε, τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και από το πρόγραμμα για την ανάκαμψη και από το πρόγραμμα εμπορίας ρήπων όπως επίσης και από τη χρήση υπαρχόντων μέσων όπως ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την δομή της επένδυσης που απαιτείται για τις πρωτοβουλίες οι οποίες ε, έχουν ήδη προταθεί. Η δομή είναι δομή συνεργατική ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αυτό θα ποικίλει βέβαια ανάλογα με το πρόγραμμα λόγω ακριβώς της εμπλοκής και της συμμετοχής της αγοράς στις διαφορετικές τεχνολογικές παρεμβάσεις. Οι προτάσεις πάντως τις οποίες κάνουμε είναι σοβαρές προτάσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εν γνώση των προβλημάτων τη συζήτηση για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. Ένα επιπλέον στοιχείο να προσθέσω ξεκινάμε με όλες τις πρωτοβουλίες φέτος εκτός από μία, τις έξυπνες πόλεις, τα smart cities. Με αυτήν θα ξεκινήσουμε το επόμενο έτος. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτά τα οποία συζητάμε τώρα δεν έχουν ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο βέβαια έρευνας. Και μάλιστα στο ερευνητικό κομμάτι οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει και πριν από αρκετό καιρό και όχι μόνο φέτος. Ένα τελευταίο στοιχείο. Προσπαθούμε να εργαστούμε σωστά σε κοινοτικό επίπεδο. Ξέρετε ότι εγώ έχω δώσει μάχες για την ευρωπαϊκή έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το 5% των ερευνητικών επενδύσεων, των επενδύσεων στην έρευνα, καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις με τα εθνικά επίπεδα. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα έχουμε συγκεκριμένους στόχους πετύχει. Τα χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να συνδυαστούν με τα χρήματα που διαθέτουν οι διάφορες χώρες. Τα προγράμματα τα κοινά τα οποία έχουμε προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και θα γίνουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποτιμήσετε αυτά τα οποία προσπαθούμε να πετύχουμε. Μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αφ' αυτού και θα υπάρξει συγκεκριμένος δημοσιονομικός κανονισμός ο οποίος θα έρθει προς συζήτηση για την κατανομή της ανάληψης των κινδύνων για να ε, διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό. Είμαστε λοιπόν πίσω από μία από τις ε, ουσιαστικά μείζονες ε, εξελίξεις στην Ευρώπη. Έχουμε τη συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ενέργεια η οποία έχει δραστηριοποιηθεί. Έχουμε τα καλύτερα ε, ερευνητικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στα, στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Και το τελικό μου μήνυμα είναι ότι είναι καθήκον όλων